αγαπητό Επίτροπο, να μην λογοκρίνετε τα λόγια μου παρακαλώ, να λέτε όχι απλά τον Κύριο, αλλά να λέτε τον αγαπητό Κύριο, γιατί το λέω σκοπίμως και ηθελημένα και θέλω να το λέτε και αυτό. Αυτά είχα να πω. Καληνύχτα σε όλες και όλους. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9.